La seduta è aperta. Κυρίσω την έναρξη της συνόδου, λέει ο πρόεδρος. Κύριε Φερβόστατ, παρακαλώ. Καθίστε. La semaine dernière. Την περασμένη εβδομάδα ναι, θλίψη μάθαμε